τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, όταν ε, ο εκλεγμένος πρόεδρος Γιούνκερ μου ανέθεσε αυτό το χαρτοφυλάκιο, είχε την ευγένεια να πει ότι ομιλώ την γλώσσα του Σέξπιρ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρξω σαφής στην μετρική μου γλώσσα, αλλά πάνω απ' όλα ήθελα στη γλώσσα του Μολιέρου, ή τέλο πάντων στη δική μου εκδοχή της γλώσσας του Μολιέρου, να σας, να σας ευχαριστήσω που με τιμήσατε με την ε, σημερινή πρόσκληση. Ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που εσείς, πολλοί από εσάς, ήδη μου διαθέσατε πριν από την ακρόαση. Σήμερα θέλω να απαντήσω στις εξής τρεις βασικές ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί θέλω αυτή τη θέση και δεύτερον, ποια είναι η εμπειρία που μπορώ να προσφέρω στις αρμοδιότητες που θα αναλάβω. Τρίτον, πώς θα προσεγγίσω το καθήκον μου, ένα λειτουργήμα που είναι τόσο σημαντικό για τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη. Οπότε και τόσο σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί θέλω αυτή τη δουλειά λοιπόν. Γιατί θα ήθελα να διαδραματίσω το ρόλο μου αποκρινόμενος σε δύο βασικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Την πρόκληση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Ευρώπη μεταξύ των πολιτών και την πρόκληση του να έχουμε και πάλι θέσεις εργασίας και ανάπτυξης στις οικονομίες μας. Προσωπικά επειδή θέλω η Βρετανία να είναι μέρος και μέλος μιας επιτυχημένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είχε λογική και νόημα για την Βρετανία, το ίδιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γενιά των γονιών μου πήγε στον πόλεμο και πολέμησε. Η δική μου γενιά μεγάλωσε σε μια χωρισμένη Ευρώπη, μια κατακαιρματισμένη Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας την απειλή της πυρηνικής εξόντωσης. Όταν, ε, όταν έπεσε το σιδηρούν παραπέτασμα Πού στράφηκαν οι νέες δημοκρατίες που αναδύθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε, είχαμε λοιπόν κάθε λόγο να αποκριθούμε σε αυτήν την ε, έκκληση. Ναι λοιπόν, θέλω να δουλέψω για το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και θέλω η χώρα μου να παραμείνει μέρος μιας ένωσης 500 εκατομμυρίων πολιτών με κοινέ αξίες που ε, συνυπάρχουν, εργάζονται μαζί, εμπορεύονται και συναλλάσσονται μεταξύ τους και αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις από κοινού. Εγώ τώρα ποιο είμαι και τι θα προσφέρω σε αυτή τη δουλειά εφόσον ε, εγκριθώ. Είμαι γιο ενό μικρού επιχειρηματία και μια δασκάλα. Έχω δουλέψει τη μισή μου ζωή στην κυβέρνηση και την άλλη μισή στον επιχειρηματικό κλάδο. Ξεκίνησα ω σύμβουλο του Κένεθ Κλάρκ και του Τζον Μέιντζορ τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Μετά από αυτό ίδρυσα τη δική μου εταιρεία, οπότε γνωρίζω ποιε είναι οι προκλήσει του να προσπαθεί κανεί να δημιουργήσει μια μικρή εταιρεία σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πριν από τέσσερα χρόνια άφησα αυτό το χώρο και ξεκίνησα να εργάζομαι στην Βρετανική κυβέρνηση ως υπουργό. Ανέκαθεν έχω ε, εγκαταλείψει όλε μου τι μετοχέ, δεν έχω καμία μετοχή στη διάθεσή μου, δεν είμαι μέλο κανενό διοικητικού συμβουλίου, οπότε δεν πιστεύω ότι στην περίπτωση μου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Το 2010 ανέλαβα υπουργό παιδεία και ανέλαβα τι μεγαλύτερε μεταρρυθμίσει στην παιδεία εδώ και μία γενιά. Έπειτα ήμουν μέλος της Βρετανικής κυβέρνησης και ε, ασχολήθηκα με την... Ε, και φρόντισα ο, ο κυβερνητικός συνασπισμός να ηγήθηκαν του κυβερνητικού συνασπισμού στη Βουλή των Λόρδων. Ε, η Βουλή των Λόρδων ασχολείται με την τροποποίηση και τροπολογία της νομοθεσίας και με τον ειδικό δημοκρατικό έλεγχο. Υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες εκεί, κανένα κόμμα δεν έχει την πλειοψηφία, το μεγαλύτερο κόμμα έχει μόλι 28% των ψήφων, οπότε ο μόνος τρόπος να προοδεύσει κανείς είναι να υπάρχει συνένεση και να, ξεπερνά, να ξεπερνώνται οι κομματικές γραμμές. Έτσι λοιπόν μπόρεσε να ε, φέρω μια περίπλοκη μεταρρύθμιση σε ένα πολύπλοκο πολιτικό περιβάλλον. Νομίζω ότι έχω δώσει ε, την, ε, αποδεικτικά στοιχεία ότι καταφέρνω να επιτύχω συνένεση και καταλαβαίνω από αυτήν την σκοπιά το θέμα των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης. Πώς θα αναλάβω τώρα το καθήκον αυτό που μου αναθέτει ο κύριος ε, Γιούνκερ. Θα συνεργαστώ με τον Γιέρκη Κατάιναν, τον Βάλτη Ντομπρόφκες και τον Πιέρ Μοσκοβισή και άλλους ε, ε, συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα συνεχίσω αυτά που έκαναν ο Μισελ Μπαρνιέ, αυτή η Επιτροπή του Κοινοβουλίου και θα φροντίσω να υπάρχει μια εύρυθμη, ε, ένας εύρυθμος κλάδος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που θα ε, εργάζεται προς το συμφέρον όλων, όχι των λίγων. Θέλουμε να είναι ισχυρό το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, κάτι που προσπαθήσαμε να το προστατεύσουμε και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι χώρος τιμής που πρέπει να αποταθεί στον ε, προκάτοχό μου. Ένα από τα βασικά στοιχεία της ε, εργασίας μας θα είναι η Τραπεζική Ένωση με, το κοινό, με τους κοινούς κανόνες και για τα 28 κράτη-μέλη. Εφόσον εγκριθώ θα φροντίσω αυτό το πάζλ να αρχίσει να λειτουργεί ώστε να υπάρχει σταθερότητα για το τραπεζικό μας σύστημα. Κάτι που όλοι επιθυμούμε. Ναι, προέρχομαι από μια χώρα εκτός της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά η πρόσφατη κρίση μας έδειξε πόσο αλληλένδετα είναι τα συμφέροντα των 28 κρατών μελών. Μια ισχυρή τραπεζική ένωση είναι σημαντική για όλους μας και θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να γίνει αυτό μια εμβληματική κίνηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στους καιρούς πρώτης κρίσης. Δεν μπορούμε πλέον να αναλαμβάνουμε μεγάλους κινδύνους που μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη θέση εργασία και το βιωτικό επίπεδο πολλών από τους πολίτες μας. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στον καιρό που οι τράπεζες έπρεπε να σώζονται εις βάρος των φορολογουμένων. Νομίζω όμω ότι όλοι συμφωνούμε για τα ερχόμενα χρόνια ότι χρειαζόμαστε νέα κίνητρα για τι θέσει εργασία και την ανάπτυξη. Πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε για του νέου κινδύνου που αναδύονται στο σύστημά μα. Όμω δεν πρέπει να φανταστούμε ότι θα χρειαστεί η ίδια νομοθεσία όπω την ε, προηγούμενη πενταετία για το ερχόμενο διάστημα. Η καλή νομοθεσία θα πρέπει να μα προσφέρει σταθερότητα αλλά και ε, αυστηρότητα. Ταυτόχρονα, εάν να παρουσιαστούν στοιχεία που δείχνουν ότι δεν έχουμε πετύχει το σωστό σημείο ισορροπία, θα πρέπει να κάνουμε τι απαραίτητε προσαρμογέ. Υπάρχουν τομεί όπου ενδεχομένω θα εντοπίσουμε ελλείψει. Τομεί όπου θα δούμε ότι πρέπει μερικά πράγματα στι λεπτομέρειέ του να προσαρμοστούν, ώστε να γίνουν οι ροέ των επενδύσεων πιο απλέ. Αυτή είναι η πρόκληση που βρίσκεται στην καρδιά τη Ένωση των Κεφαλαιοχικών Αγορών. Το πώ θα αυξήσουμε τι επενδύσει, ιδίω προ τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, ενώ θα συνεχίσει να αποτελεσματική νομοθεσία είναι ένα βασικό θέμα που θα μας απασχολήσει. Μέσα σε αυτήν την γενικότερη προσέγγιση έχω θέσει στον εαυτό μου τέσσερις βασικές προτεραιότητες. Πρώτον, να υλοποιηθούν όσα ήδη συμφωνήθηκαν. Αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ σοβαρό καθήκον. Η κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικέ πράξει είναι περίπου 400 ξεχωριστά μέτρα από το MIFID 2 στην Τραπεζική Ένωση, στο Solvency 2 και στο CRD. Σε κάθε τι που κάνουμε θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μια δίκαιη και ανοιχτή διαφανή διαδικασία. Σε συνεργασία με εσά και το Συμβούλιο. Έπειτα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλε βασικέ πηγέ κινδύνου. Με την προώθηση προτάσεων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, όπω ε, τα ταμεία για τι ε, χρηματοπιστωτικέ αγορέ, την συγκριτική αξιολόγηση και τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των αναδυόμενων κινδύνων, επειδή κάποιε φορέ δεν υπάρχει ένα αρκετά αποτελεσματικό σύστημα επαναγορά για, για τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τρίτον, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει σαφή υλοποίηση και κάλυψη των ελλείψεων που μπορεί να απειλούν την χρηματοπιστωτική μα και δημοσιονομική σταθερότητα. Θα συνεργαστούμε και με τι υπόλοιπε χώρε του G20 και ιδιαίτερω θα θέλαμε μεγαλύτερη ρυθμιστική συνεργασία με τι ΗΠΑ. Κατά τέταρτον, θα υποβάλω προτάσει για να αναπτυχθεί η Ένωση των Κυβερνητικών Αγορών. Αυτό είναι ένα εγχείρημα που αφορά και τα 28 κράτη-μέλη. Ο στόχο είναι σαφής Θέλουμε να απελευθερωθεί το κεφάλαιο που περιβάλλει την Ευρώπη και αυτή τη στιγμή έχει παγώσει και επιτέλους να εξυπηρετήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες. Θέλουμε να ε, ξεφύγουμε από την εξάρτησή μας από την χρηματοδότηση των τραπεζών και να αναπτύξουμε νέες εναλλακτικέ πηγές χρηματοδότησης. Θα πρέπει να αναλύσουμε το πρόβλημα και τους φραγμούς που υπάρχουν για την πρόοδο ενός τέτοιου εγχειρήματος ω τώρα. Αλλά νομίζω ότι ήδη εντοπίζουμε κάποιους πιθανούς τομείς όπου θα πρέπει να ε, στρέψουμε ήδη την προσοχή όπως ε, την ε, υψηλή την υψηλή ε, πληροφόρηση για το, την πιστοληπτική ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μια συμφωνία για, τα, για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τα ταμεία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα ωφέλη που μπορεί να δώσει η ενιαία αγορά απευθείας στους πολίτες. Ε, Όντω και δικαίω τα τελευταία πέντε χρόνια επικεντρωθήκαμε στι μεγάλε διευθυντικέ και θεσμικέ μεταρρυθμίσει που χρειάζονταν. Την ερχόμενη πενταετία πιστεύω ότι μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μα προ μια άλλη κατεύθυνση και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώ θα έχουμε μια καλύτερη αγορά για ασφαλεί, διαφανεί και κερδοφόρε ε, πωλήσει ε, λιανική. Ε, ήδη στο σώμα αυτό βλέπουμε ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στα συμφέροντα των καταναλωτών και θα σας στηρίξω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια τα ερχόμενα χρόνια. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις ψηφιακές και ηλεκτρονικές πληρωμές που μπορεί να δώσουν μεγάλα ωφέλη στους καταναλωτές από την άποψη του κόστους και να διευκολύνουν τη χρήση αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ασφαλείς και σωστά ρυθμισμένες και αυτές. Υπάρχει όμως ένα βασικό θέμα που ξεπερνά όλα τα άλλα και αυτό νομίζω ότι είναι η διαφάνεια είναι καθοριστική σημασία από την άποψη των όσων απαιτούμε να κάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα πρέπει να γνωρίζουν τι κινδύνου αναλαμβάνουν και να εξηγούν του κινδύνου αυτού και στου ε, πελάτε του. Οι εποπτέ θα πρέπει να το γνωρίζουν επίση. Οι περισσότεροι κανόνε που έχετε θεσπίσει κι εσεί, όλοι ε, προβλέπουν αυστηρότατε προποθέσει και απαιτήσει διαφάνεια. Και αυτό είναι πολύ σωστό για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των πολιτών Πώς θα συνεργαστώ τώρα μαζί σας εφόσον ε, με εγκρίνετε. Ε, κατά πρώτον, η διαφάνεια θα είναι ένα βασικό στοιχείο στη συνεργασία μας. Θα υπάρχει ανοιχτός διάλογος με αυτή την Επιτροπή ανα πάσα στιγμή και θα σας ενημερώνω και για τις συναντήσεις μου για να ε, μπορέσω να φέρω εις πέρα στο καθήκον μου. Θα μιλήσω με μια σειρά από ανθρώπους που πιστεύω ότι θα πρέπει να του συναντήσω, γιατί δεν μπορεί κανείς να χαράζει πολιτική σε ένα κενό αλλά θα ακολουθήσω και τις ε, ε, προδιαγραφές της, τα πρότυπα του προκατόχου μου, ώστε να ενημερώνω και για εξωτερικές συναντήσεις, το ίδιο και οι συνεργάτες μου. Αυτό νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό και για εσά και για να έχουμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη μεταξύ μα. Στο Στρασβούργο τη προάλλη συναντήθηκα με τον Μισελ Μπανιέ και ζήτησα τι συμβουλέ του. Είχε πολλέ χρήσιμε μικροσυμβουλέ να μου δώσει, αλλά ήταν ένα το σημαντικότερο από αυτά που μου είπε. Πάντοτε να θυμάσαι, είπε, τη σημασία τη σχέση σου με αυτό το σώμα, με το κοινοβούλιο. Αυτήν την συμβουλή πραγματικά την έλαβα πολύ σοβαρά υπόψη μου και είναι μια συμβουλή την οποία θα φροντίσω να ακολουθήσω. Ξέρω ότι ο πρόεδρο Γιούνκερ μου έχει αναθέσει μια μεγάλη ευθύνη ζητώντα μου να αναλάβω αυτό το χαρτοφυλάκιο. Εφόσον λάβω την έγκρισή σα, θα είμαι ο Ευρωπαίο Επίτροπο που προασπίζεται το γενικό συμφέρον. Ένα Ευρωπαίο Επίτροπο που θα εργάζεται προ όφελο και των 28 κρατών μελών. Ένα Ευρωπαίο Επίτροπο που ποτέ δεν θα ξεχνά ότι πρέπει να λογοδοτήσει τα άμεσα εκλεγμένα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ.